θέμα στην ημερήσια διάταξη επίσης ε, ένα θέμα στο οποίο θα κάνει δήλωση η πατή εκπρόσωπος ε, της Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και το θέμα είναι η απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στην Δυτική Όχθη. Και πάλι στρέφω προς το Συμβούλιο. Κυρία Μαρκουλή, μπορείτε να κάνετε την ε, δήλωσή σας. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, όπως γνωρίζετε την Δευτέρα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων εξέδωσε συμπεράσματα σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Κανείς δεν αμφιβάλλει για την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί αυτού του κρισίμου ζητήματος. Η θέση είναι σαφής και θα προϋποθεί και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αλλά έχουμε και την δήλωση της 29ης Νοεμβρίου. Η επανεκκίνηση των απευθεία διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών χωρί καθυστέρηση ή προποθέσει είναι αυτό το οποίο επιδιώκει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σαφέ ότι θα περιθούν προ τούτο σαφή γενναία βήματα και από τι δύο πλευρέ. Όμως, σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι απευθείας ουσιαστικές συνομιλίες είναι απολύτως απαραίτητες για να επιτευχθεί μια βιώσιμη διαρκής λύση στην διαμάχη Παλαιστινίων Ισραήλ. Χρειάζονται σαφείς παράμετροι εν ώψη της διαπραγμάτευσης για να εξασφαλιστεί επιτυχές αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διερεθειμένη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένε Πολιτείες και άλλους διεθνείς παράγοντες, όπως με την τετραμερή, με κοινό σκοπό ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη ειρήνευσης το 2013. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί επίσης με όλες εκείνες τις πλευρές που θέλουν να επιτύχουν ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία στην περιοχή. Η Ελληνική Πρωτοβουλία συγκεκριμένα παρέχει υποστήριξη για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Όλες οι πλευρές πρέπει να αποφύγουν ενέργειες που θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη ή την βιωσιμότητα της λύσης των δύο κρατών. Από την διακήρυξη της Βενετίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι οι επικισμοί είναι παράνομη βάση του διεθνούς δικαίου και αποτελούν εμπόδιο στην ειρήνη. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι τη Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την βαθιά της ανησυχία και σαφή αντίδραση στα Ισραηλινά σχέδια. Μετά και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών στις 29 Νοεμβρίου. Σχετικά δηλαδή με την επέκταση των των οικισμών μεταξύ άλλων και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το σχέδιο αυτό, εάν υλοποιηθεί, θα υπονομεύσει σοβαρότατα τις πιθανότητες ειρηνικής επίλυσης της διαμάχης. Υπονομεύοντας δηλαδή τις προπτικές δημιουργίας ενός συνεκτικού Παλαιστινιακού κράτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι θα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις καθώς και τις εν γέννη επιπτώσεις τους και θα αναλάβει αναλόγως δράση. Με άλλα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν ποτέ σαφέστερη. Το ίδιο έκανε και την Δευτέρα. Η υλοποίηση αυτών των σχεδίων όχι μόνο θα έχει επιπτώσεις στις προοπτικές δημιουργίες Παλαιστινιακού κράτους, επιπλέον θα έχει επιπτώσεις Στι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Με το ίδιο πνεύμα η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την δέσμευσή της να διασφαλίσει ότι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο όλες οι συμφωνίες μεταξύ του Ισραήλ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει απερίφραστα και ρητό να περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι δεν εφαρμόζονται, δεν ισχύουν στα σύνορα εκτό του Ισραήλ με τα σύνορα του 67. Επίσης επαναδιατυπώσαμε τη δεσμευσή μας να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά και αδιάλειπτα την ευρωπαϊκή νομοθεσία στις διμερείς ρυθμίσεις που αφορούν τους νέους οικισμούς. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να αποφύγει κάθε βήμα, κάθε ενέργεια που υπονομεύει την οικονομική κατάσταση της Παλαιστινιακής Αρχής. Οι σημερινές υποχρεώσεις βάσει δι του πρωτοκόλλου του Παρισιού πρέπει να γίνουν σεβαστές και ιδίως αφορά τη μεταφορά των σχετικών εσόδων στην Παλαιστινική Αρχή. Επίσης η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει να χρησιμοποιήσει, να αξιοποιήσει αποδοτικά, επικοδομητικά το νέο καθεστώς των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Έθνη και να μην αναλάβουν ενέργειες οι οποίες θα υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη και που θα απομειώσουν τις πιθανότητες επίτευξης ειρηνευτικής λύσης. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, μόλι πριν από τρει εβδομάδε συζητούσαμε τις τελευταίες εχθροπραξίε μεταξύ τη Λωρίδα της Γάζα και του Ισραήλ που κατέληξαν σε εκεχηρία λίγο αργότερα τη νύχτα εκείνη που θα θυμάστε. Η Δευτέρα ήταν μάλιστα η πρώτη ευκαιρία για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων να καταγράψει την εκεχηρία και να συζητήσει την περαιτέρω συνδρομή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε η εκεχηρία αυτή να είναι βιώσιμη. Η εκεχηρία αυτή κρατάει προς το παρόν. Έχει μεγάλη σημασία όλα τα μέρη που συνυπέγραψαν την οικηγυρία να συνεχίσουν να την τηρούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να διευκολύνει τις οικονομικές και κοινωνικές πρόοδους στην Λωρίδα της Γάζας. Επίσης, η εισαγωγή όπλων στη Λωρίδα της Γάζας πρέπει να αντιμετωπιστεί αμέσως. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα με την διερμηνία σε άλλε γλώσσε, λέει ο πρόεδρο και διακόπτει την κυρία Μαρκουλή. Ποια γλώσσα δεν ακούγεται. Γαλλικά. Πολύ ωραία. Έχουμε διερμηνία τώρα σε όλε τι γλώσσε. Με συγχωρείτε κυρία Μαρκουλή. Παρακαλώ συνεχίστε. Είχαμε μια διακοπή. Είχαμε μια διακοπή μεγάλη διάρκεια, λέει κάποιο από την αίθουσα. Αναγνωρίζουμε τις ανάγκε ασφαλείας του Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναδιατυπώνει την έκκλησή της για άμεση προσπάθεια να ανοίξουν τα σύνορα για να αποκρισταθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, εμπορευμάτων και προσώπων από και προς τη λωρίδα της Γάζας. Είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο εργαλείο για να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες των δύο μερών συμπεριλαμβανομένης της επανεργοποίησης της αποστολής EUBAM στη Ράφα. Επίσης, επαναδιατυπώσαμε τη δέσμευσή μας υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης των απειλών που αντιμετωπίζει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα σταματήσει να αντιτίθεται σε αυτούς που προωθούν την δημοκρατία και την βία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επανάληψη έχει απευθύνει έκκληση για συμφιλίωση μεταξύ των Παλαιστινίων υποστηρίζοντας τον πρόεδρο Αμπάς βάσει των αρχών της ομιλίας του, του Μαΐου του 2011. Αυτό θα αποτελέσει ουσιαστικό στοιχείο της ενότητας εν του Παλαιστινικού κράτους για να πετύχουμε εν τέλει τη λύση των δύο κρατών. Η συμφιλίωση αυτή θα έχει επίσης αμέσως επιπτώσεις στην κατάσταση στην λωρίδα της Γάζας, η οποία δεν είναι βιώσιμη και είναι απαράδεκτη όσο η λωρίδα της Γάζας παραμένει αποκομμένη από την εθνική Όχθη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προσβλέπω στην υπερψήφιση του σχετικού ψηφίσματος αύριο. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Εξ του ΕΛΚ, ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Έχετε δυόμιση λεπτά κύριε Γκάλερ στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαπιστώνουμε πως αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει το πάνω χέρι. Εμείς ε, επιμένουμε στην βάση των διεθνών συμφωνιών, δηλαδή μια λύση δύο κρατών. Βεβαίω η λύση της σύγκρουσης αυτής δεν θα ωφελήσει μόνο τους εμπλεκόμενους, ε, θα ωφελήσει άμεσα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό δεν πρέπει μόνο να αντιδράμε ή να κάνουμε δηλώσει. Πρέπει πρώτα απ' όλα να κατονομάσουμε όσου εμποδίζουν την ενεργειακή διαδικασία. Δηλαδή από πλευρά Παλαιστινίων το, τα πλήγματα κατά του Ισραήλ από τη Λόριδα του Σικάζας καθώς και οι δηλώσει ε, του πρόεδρου τη Χαμάς να ότι θα σβήσει το Ισραήλ από τον χάρτη. Επίσης θα πρέπει πράγματι να αναγνωρίσουμε πως ε, ναι βεβαίως έχει το δικαίωμα να υφίσταται το Ισραήλ ως ένα Ιουδαϊκό κράτος αλλά βεβαίως βλέπουμε πως η κυβέρνησή του ε, δεν ε, ακολουθεί και δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό, δεν ακολουθεί τις μεύσεις και δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για την ειρήνη. Όλοι οι οικισμοί είναι παράνομοι, αυτή είναι η νομική και πολιτική μας πεποίθηση, γι' αυτό ζητάμε μόνιμη και ε, άμεση, άμεσο σταμάτημα αυτών των ε, δραστηριοτήτων. Επίσης σχετίζω αυτό το οποίο είπατε για την απόδοση των ε, δασμολογικών εσόδων. Και βεβαίω θα πρέπει να δούμε ποια μέτρα μπορούμε να αναμένουμε από την Παλαιστινική κυβέρνηση μέχρι ποια προθεσμία και η Ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να αναρωτηθεί το πού οφείλεται το ε, ότι υπήρχε μόνο ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταψήφισε την αναγνώριση της ε, Παλαιστίνης. Δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η οποία άλλαξε. Επίσης θα πρέπει να μην υπάρχει ε, να μην εκμεταλλεύονται ιδρύματα στα κατεχόμενα την συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα πανεπιστήμιο στο Άριελ, παραδείγματο χάρη. Αυτά πρέπει να τα λάβει υπόψη του Ισραήλ και μάλιστα Σε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Θέλετε να απαντήσετε μια ερώτηση με την μπλε κάρτα. Κύριε Μέρφυ, έχετε το λόγο. Thank you. Could I ask the member... Ευχαριστώ να ρωτήσω τον κύριο συνάδελφο εάν υπερψήφισε την αναβάθμιση των υπουργικών σχέσεων με το Ισραήλ πριν από δύο μήνες. Θεωρεί πως μόνο η κριτική φτάνει ή πρέπει να κάνει και κάτι το Κοινοβούλιο έτσι για αλλαγή. Όσον αφορά την συμφωνία αυτή, εγώ δεν τη θεώρησα αναβάθμιση, ήταν συνέχεια υφισταμένων πραγμάτων. Δεν ήταν καμία αναβάθμιση και την υπερψήφισα. Και συμφωνώ το Κοινοβούλιο δεν είναι εκτελεστική εξουσία. Απευθύνω έκκληση στο Συμβούλιο, την Κομισιόν, τα κράτη-μέλη να δράσουν ανάλογα με αυτά τα οποία είπα, να ορίσουν στόχους, χρονοδιάγραμμα, συγκεκριμένες προτάσεις και αν δεν γίνει τίποτα να αντιδράσουμε. Είτε προς τους Παλαιστινίους είτε προς τους Ισραηλινούς. Ε, Πραγματικά με δυσαρεστεί το ότι η τωρινή κυβέρνηση δεν βλέπει σωστά το μέλλον της ε, χώρας της και είναι σκληρή η δήλωσή μου και με θλίψη μου την κάνω. Ε, ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι η κυρία Γκόμες ο επικισμός στη Δυτική Όχθη είναι κάτι που έχει οδηγήσει σε μεγάλες αντιδράσεις. Μιλάμε για 3.000 νέες κατοικίες, κάτι τα οποία είναι μια μεγάλη πρόκληση για την Παλαιστίνη και μια μεγάλη ήττα που επιβάλλει στον εαυτό του το Ισραήλ. Γιατί ο μόνος τρόπος για να φτάσουμε στην ειρήνη είναι να υπάρχει ειρηνική συνύπαρξη με ένα κράτος της ε, Παλαιστίνης το οποίο θα είναι πλήρως λειτουργικό και βιώσιμο. Θα πρέπει να δράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και οι παράνομοι επικισμοί θα πρέπει να σταματήσουν και να υπάρξουν επιπτώσεις στις εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Επίσης και προς την Χαμάς θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποστείλει ένα σαφές μήνυμα. Το κράτος του Ισραήλ είναι υπαρκτό και κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξή του. Τι θα γίνει όμως με την δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους που θα ζει δίπλα-δίπλα με το Ισραήλ ειρηνικά. Εξ ονόματος των φιλελευθέρων κυρία Νέης. Κύριε... Κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, όταν ξεκινήσαμε να προετοιμάζουμε τα διάφορα σχέδια του σημερινού ψηφίσματος, δεν ξέραμε ακόμα τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Δευτέρας. Παρ' όλα αυτά, όταν συγκρίνει κανείς το αρχικό κείμενο και το κείμενο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, βλέπει πάρα πολλά α, στοιχεία παραλληλισμού στην προσέγγιση μας. Βεβαίως, λυπούμεθα για τις ανακοινώσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης, για την οικοδόμηση περαιτέρω οικισμών στην περιοχή ε1 η οποία αν εφαρμοστεί ποτέ το ειρηνευτικό σχέδιο αν εφαρμοστούν ποτέ αυτά τα σχέδια κατ' ουσίαν θα καταστήσουν ε, αδύνατον ένα εδαφικά συνεχές Παλαιστινιακό κράτος και συνεχίζουν να κατακρατούν και δασμούς ε, και οι δύο αυτές ανακοινώσεις ε, γίναν μέρες μετά την ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μου φαίνεται πως με τις ανακοινώσεις αυτές η Ισραηλινή κυβέρνηση υπονομεύει την νομιμότητα του Μαχμούντα Μπάς και εξ αντανακλάσεως αυτή η υπονόμευση δεν μπορεί παρά να ενισχύσει την Χαμάς η οποία κατά την ε, άποψη του Ισραήλ ε, είναι μια συμπεριφορά παράδοξη καλωσορίσαμε και καλωσορίζω τα συμπεράσματα, όπως είπα, του Συμβουλίου Υπουργών και θεωρώ πως η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος και η ομάδα της έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο με το να καταλήξουν σε αυτά τα συμπεράσματα δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αυτά τα συμπεράσματα έχουν εγκριθεί ομόφωνα και από το 27 κράτη-μέλη και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτεί η Ισραηλινή κυβέρνηση. Αναλύοντας προσεκτικά την ε, ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ. Όπως είπε ο κ. Γκάλέ. είναι σημαντικό το ότι μόνο ένα κράτος μέλος συντάχθηκε με το Ισραήλ και τα άλλα είτε υπερψήφισαν την πρόταση της Παλαιστίνης είτε απήχαν. Εάν η κυβέρνηση του Ισραήλ συνεχίσει να δρά με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί τελείως απομονωμένη. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί θα γίνει πιο δύσκολη να ζητήσει η μόνιμης λύσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εξονόμου των Πρασίνων και της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας. Το λόγο έχει η κυρία Πράντνερ για ένα μισή λεπτό. Σας καλωσορίσω κυρία Υπουργέ. Η επέκταση των οικισμών στην ζώνη ε1 είναι κάτι το απαράδεκτο, γιατί έτσι δεν, είναι, δεν γίνεται βιώσιμο το Ισραηλινό, κράτος. Χτες το πρωί έγινε μία επίθεση στην Ένωση των Γυναικών και σε άλλες ΜΚΟ Πολλές ΜΚΟ τις υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι αυτό αποτελεί απειλή στην ειρηνευτική διαδικασία της περιοχής και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν προωθούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε καμία από τις δύο χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ότι στο τελευταίο ε, Συμβούλιο Σύνδεσης με το Ισραήλ να προωθηθούν 60 νέες δραστηριότητες. Προτείνω να γίνει πάγωμα αυτών των δραστηριοτήτων ε, καταδεικνύοντας έτσι ότι δεν δεχόμαστε την, ε, την στάση του Ισραήλ και τις πρόσφατες πράξεις τους. Επίσης, θεωρώ ότι θα πρέπει να δείξουμε μέσω, ε, μέσω του πρέσβη μας ότι ότι δεν δεχόμαστε τους παράνομους επικισμούς. Δεν πρόκειται για κάτι που αφορά το Ισραήλ, δηλαδή δεν αντιτιθέμεθα στο κράτος του Ισραήλ, αλλά στην παρούσα κυβέρνηση. Εξ των συντηρητικών, ο κύριος Τάνοκ. Κατανοώ ησυχίες των Ισραηλινών και Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και θυμός από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Βλέπουμε ότι έχει παραβιαστεί η συνθήκη του Όσλο όμως του 1993. Η ομάδα μου έχει αντιταχθεί στις επεκτάσεις και στις ε, δημιουργίες νέων επικισμών και οι τελευταίες Ισραηλινές ανακοινώσεις δεν βοηθούν το Ισραήλ. Όμως ο διάβλος ε1 είναι σε φάση προγραμματισμού και η κυβέρνηση δεν μιλά για επικείμενες εργασίες, απλώς δεν καταβάλλονται ε, χρήματα στην Παλαιστινιακή Αρχή για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα λειτουργικά του έξοδα. Η κατάσταση θα πρέπει να αποκλιμακωθεί, θα πρέπει όλοι να δείξουν ταπεινοφροσύνη και σύνεση και να γυρίσουν στο, στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων για να υπάρξει λύση με δημιουργία δύο κρατών, με ύπαρξη δύο κρατών. Στη συμφωνία του Όσλο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ελέγχθη ότι το θέμα των επικισμών έπρεπε να επιληθεί μετά από ε, διμερείς. Οι επικισμοί δεν είναι η βασική, ο βασικός λόγος σύραξης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η επιθετική πολιτική του Ισραήλ άρχισε 50 χρόνια πριν στη Δυτική Όχθη. Και οι Παλαιστινιακές αρχές και οι τρομοκράτες της Χαμάς δεν δέχονται την ε, νομιμότητα του κράτους του Ισραήλ ως εβραϊκό κράτος. Άρα το θέμα δεν είναι καθαρά εδαφικό, αλλά είναι και θέμα νομιμότητας και δεν θα φτάσουμε σε ε, βιώσιμη λύση αν δεν το δεχτούμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να διοργανηθεί μία ακρόαση για να ακούσουμε εμπειρογνώμονες και νόμα μαθής και από τις δύο πλευρές και για να φτάσουμε σε καλύτερη πληροφόρηση έχοντας ένα ιστορικό και νομικό υπόβαθρο του ζητήματος. Ευχαριστώ πολύ. Εξ της ε, ΓΚΟΕ, ο κύριος Λεγιαρίκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Παλαιστινιακή Αρχή και ο Μαχμούτ Αμπάς χρησιμοποιούν τη διεθνή διπλωματία. Η Ισραηλική κυβέρνηση όμως ε, δέχθηκε τη βία και παραβίασε σκοπίμως τις διεθνείς συνθήκες. Εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ώστε μια κυβέρνηση να τηρεί τέτοια στάση. Πρόκειται για μονομερή σχέδια κατά, του, ε, κατά της ε, συνέλευσης, της Συνέλευσης του, των Ηνωμένων Εθνών που δέχτηκε την Παλαιστίνη ως χώρα παρατηρητή. Θα πρέπει να επικρατήσει το διεθνές δίκαιο και να μην ε, δεχόμαστε ώστε το Ισραήλ να παρακρατεί τους φόρους που πρέπει να αποδοθούν στην Παλαιστινιακή Αρχή και να συνεχίσει τους επικισμούς. Γίνεται λόγος για τη ζώνη ε1. Όμως έτσι θα αποτραπεί η δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους Εάν ε, κρατηθεί αυτή η ζώνη γι' αυτό, η Δυτική Όχθη και η Ιερουσαλήμ αποτελούν την Παλαιστίνη. Το Ισραήλ φέρει μεγάλη ευθύνη, διότι προσυπογράφοντας την ε, συνθήκη της Γενέβης το 51 και το άρθρο 41 που δεν θέχεται τους επικισμούς μετά από ε, σύραξη μας δείχνει ότι δεν υπάρχει διεθνής νομιμότητα. Το άρθρο 41 αναφέρει ότι δεν μπορεί να ε, γίνει ε, μεταφορά πληθυσμών, βίαιη μεταφορά πληθυσμών και αυτό το προσυπέγραψε και το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά υποστηρίζει την κοινή πρόταση ψηφίσματος κατά της ε, βίας του Ισραήλ, που θέλει να επιβάλλει το Ισραήλ. Ευχαριστώ. Ναι. Περνάμε στους επόμενους ομιλητές. Ο κύριος Πέτερη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ειρήνη στην Μέση Ανατολή έχει στρατηγική σημασία για την Ευρώπη, τον κόσμο και για τον διάλογο, τον πολιτισμό και πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτικής μας. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ζει με ασφάλεια και Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας λέει μάλιστα πως ε, ανήκει, προς το, στο εθνικό συμφέρον της Γερμανίας η υπεράσπιση του Ισραήλ. Επίσης, είναι λυπηρό αυτό το οποίο είπε και της, της Χαμάς ότι δεν θέλει να αναγνωρίσει το Ισραήλ. Αυτή είναι η μία πλευρά, αλλά και η Παλαιστίνη έχει το δικαίωμα να ζει μέσα σε ασφαλή σύνορα. Γι' αυτό πραγματικά μας θλίβει όταν το Ισραήλ ανακοινώνει πως θέλει να χτίσει 300 νέες κατοικίες. Θέλει να ιδιοποιηθεί κάτι το οποίο δεν του ανήκει και η αιτιολόγηση είναι εκπληκτική γιατί γίνεται με την λογική της τιμωρίας γιατί ήθελε η Παλαιστίνη να αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και ε, υπήρξε μια μεγάλη πλειοψηφία υπέρ του να γίνει κράτος παρατηρητής. Οπότε το Ισραήλ πλέον ε, είναι σε αντίθεση με τη μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών του ΟΗΕ. Εάν οικοδομηθούν αυτές οι κατοικίες δεν θα είναι δυνατή πλέον η λύση των δύο κρατών και το Ισραήλ ακολουθεί έναν σκοτεινό δρόμο. Εμείς οι φίλοι του Ισραήλ πρέπει να πούμε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι η αλήθεια. Η φιλία δεν είναι να λέμε αυτά τα οποία θέλει να ακούει ο άλλος, αλλά να πούμε πως ο άλλος ακολουθεί λανθασμένο δρόμο. Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει να επιτρέψει να εμποδιστεί η λύση των δύο κρατών μέσω της οικοδόμησης οικισμών. Και όταν ο... συκοφαντείται ο πρόεδρος ε, Αμπάς ε, και ο Υπουργός Εσωτερικών Φαγιάντ πρέπει να το απορρίπτουμε. Είναι άνθρωποι που θέλουν την ειρήνη και ευχαριστώ την ε, κυρία Υπουργό για το ότι αναγνώρισε ειδικά τον ρόλο του Πρόεδρου Αμπάς. Θέλουμε να υπάρξει συμφιλίωση μεταξύ Χαμάς και Φατάχ. Είναι σημαντικό αυτό για να υπάρξει μια λύση και ζητάμε από Ισραήλ και Παλαιστίνη να ακολουθήσουν την οδό των διαπραγματεύσεων. Είμαστε υπέρ της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη και το ότι είναι δυνατή η ειρήνη το δείχνει και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το οποίο δόθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση χτες. Θεωρούμε λοιπόν πως και εκεί πέρα είναι η ειρήνη και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Ε, ευχαριστώ. Η κυρία Κοστέλα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, Συζητήσαμε πριν από ένα μήνα την κατάσταση στην Γάζα. Με ανακούφιση μάθαμε για την εκεχηρία. Εκφράσαμε υποστήριξη στο Παλαιστινιακό αίτημα για να αναγνωριστούν ως παρατηρητές στα έθνια. Έθνη. Πιστέψαμε ότι αυτό θα συμμετοδοτούσε και την επανέναρξη των συνομιλιών. Όμως τα Ισραηλινά αντίπεινα με τη μορφή τριών χιλιάδων οικισμών αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στην ειρήνη. Και αυτό το καταδικάζουμε. Το σχέδιο αυτό υπονομεύει μια για πάντα την λύση των δύο κρατών. Η παρακράτηση των φόρων από την Παλαιστινιακή Αρχή επίσης υπονομεύει την θέση του Προεδρού Αμπάς, ο οποίος είναι υπέρ μιας ειρηνικής λύσης. Χρειάζεται, είναι σαφές, άμεσο πάγωμα της επέκτασης των οικισμών, καταστροφή των οικοδομών. Πρέπει να αρθεί επίσης ο αποκλεισμό της Γάζας. Χρειαζόμαστε πρόοδο επίσης στην διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ των Παλαιστινίων, αλλά κυρίως χρειαζόμαστε επανέναρξη ανεφόρων των ειρηνευτικών συνομιλιών. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου καλούν για μέτρα και γενναία βήματα. Πρέπει να είμαστε ενεργοί, να είμαστε γενναίοι και να κινηθούμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Αλλιώς τα ωραία μας ψηφίσματα και τα ωραία λόγια θα παραμείνουν κενό γράμμα. Τα λόγια πρέπει να συνεδευτούν από πράξεις. Ευχαριστώ πολύ. Μπλε κάρτα την αποδέχεστε. Κύριε Σίνκλερ, παρακαλώ. Πρόεδρε, να συγχαρώ τη συνάδελφο για την ομιλία της, τόσο γεμάτη νόημα. Όμως θα συμφωνήσετε, ελπίζω μαζί μου, ότι ένα από τα βασικά εμπόδια στην ειρηνευτική διαδικασία είναι η άρεση της Χαμάς να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Αυτό δεν μας το είπατε. Και αυτό είναι τελικώς το πρώτο βήμα για την ειρηνευτική διαδικασία. Ε, καλό τη συνάδελφο να καλέσει την Χαμάς να αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Ευχαριστώ τη συνάδελφο για την ερώτηση. Ανέκαθεν υποστήριξε τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το δικαίωμα των Παλαιστινίων στο να αποκτήσουν το δικό τους κράτος, εννοείται ότι το ίδιο δικαίωμα έχει και το Ισραήλ εντός των συνόρων του. Ελπίζω και Καλό τους Παλαιστινίους να το λάβουν αυτό υπόψη τους. Θα φροντίσω να κάνω ό,τι μπορώ για την εσωτερική συμφιλίωση μεταξύ των Παλαιστινίων και για την επανένεξη των συνομιλιών με το Ισραήλ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Επόμενο ομιλητή, κύριε Άουκεν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο πρέπει να τονίσουμε σήμερα στο Συμβούλιο. Κάντε κάτι. Στο σημείο 3 της πολύ καλής δήλωσης της Δευτέρας αναφέρεται πως ε, πρέπει να υπάρξει ανάλογη δράση. Πολλά λόγια, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως η Ισραηλή κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρω για το τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΔΕ Υπουργός Συνδερικών χτες ε, παρομοίωσε αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το ολοκαύτωμα. Πρέπει να ζητήσει συγνώμη. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο ε, και πλέον ε, ηρωνεύονται και εμάς και το ολοκαύτωμα. Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια. Πρέπει να γίνουν πράξεις, αλλιώς ε, τα πράγματα θα στραβά. Όλοι οι Ισραηλινοί φίλοι μας μας παρακαλάνε να κινητοποιηθούμε. Τώρα υπάρχει ευκαιρία να γίνει κάτι. Σε λίγους μήνες θα έχουν χαθεί τα πάντα. Ευχαριστώ. Κύριο Σανόντεν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως η Ισραηλινή ανακοίνωση ήταν ε, λυπηρή, αλλά δεν ήταν ε, και τελείως μη αναμενόμενη μετά τη μονομερή δράση στην ε, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία αντιβαίνει πλήρως τις συμφωνίες του Όσλο. Δεν θυμάμαι επίσης κανένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου να καταδικάζει αυτή την κίνηση. Οπωσδήποτε πολλοί από εμάς εκφράσαμε την ανησυχία μας και την απογοήτευσή μας τους Ισραηλινούς ότι ε, δεν θα έπρεπε να δράσουν με τον τρόπο που έδρασαν. Γνωρίζουμε πως η κατάσταση ασφαλείας και οι εκλογικές πιέσεις οδηγούν σε δηλώσεις και πράξεις που δεν θα γίνονταν σε καιρούς πιο ήρεμους. Το εάν ε, όντως γίνουν αυτές οι κατασκευές στο ε1 που δεν νομίζω θα γίνουν, δεν είναι το βασικό θέμα. Εμένα με ανησυχούν οι γενικότερες εξελίξεις. Η Γάζα είναι ένα μέρο όπου κολλάπτεται η τρομοκρατία. Η Παλαιστίνη είναι διχασμένη, ο Μαχμούντα Μπάς δεν έχει εξουσία στην Γάζα και απουσιάζει από τι διαπραγματεύσει. Και υπάρχει βέβαια και ένα ερωτηματικό για το κατά πόσον έχει διεισδύσει και στη δυτική όχθη η Χαμάς. Και τώρα είναι ένα σύμμαχό του στην εξουσία στην Αίγυπτο, Όπω έχουμε μια λύση τριών κρατών. Και υπάρχει και η απειλή του Ιράν. Τέλος, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δράσει εκεί όπου έχει περιθώρια, δηλαδή ρεαλιστικά με τους Παλαιστινίους. Τους έχουμε δώσει 5 δισεκατομμύρια και τι έχει αποδώσει αυτή η επένδυσή μας. Πρέπει να επανέλθουν στην Τραπέζα των διαπραγματεύσεων και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Σχεδόν δύο λεπτά μιλήσατε, αλλά Έχετε ακόμη τη δυνατότητα να επανέλθετε γιατί η κυρία Άουκεντ θέλει να σας απευθύνει ένα ερώτημα. Θέλετε να απαντήσετε. Φαινόταν. Δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Είπατε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να καταδικάσει την κίνηση των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς που υπερεμεινόμεθα του κράτου δικαίου να καταδικάσουμε την κίνηση των Παλαιστινίων στα Ηνωμένα Έθνη. Και εγώ δεν πιστεύω στα αυτιά μου πολύ συχνά σε αυτό το <laughs> κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Στην περίπτωση αυτή, βεβαίω, η κίνηση των Παλαιστινίων ήταν προκλητική και μονομερής και δεν βοήθησε. Νομίζω ότι αντιτίθεται στο Όσλο. Είχαμε πει για λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Πείτε μου εσείς πώς βοηθάνε οι Παλαιστίνοι σε αυτήν την περίπτωση. Είπαμε να καθίσουμε γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και είπα ότι τώρα είναι ευκαιρία να πιέσουμε τους Παλαιστινίους να καθίσουν γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Εδώ πηγαίνουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση εντελώς. Πρόεδρος, ο επόμενος ομιλητής, κύριε Άντερσον. Ευχαριστώ. Η απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους παράνομους οικισμούς στην Δυτική Όχθη είναι ξεκάθαρα αντίπεινα κατά του Παλαιστινιακού λαού μετά την επιτυχία του στον ΟΗΕ. Η επιθετική αυτή πράξη συνεχίζει την αδιαφορία της Ισραηλινής κυβέρνησης για το διεθνές δικαίο και πρέπει να καταδικαστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Μαζί βεβαίως με την κατακράτηση 100 εκατομμυρίων δολαρίων είπα σε δασμούς που πρέπει να αποδοθούν στην Παλαιστίνη και έτσι διακινδυνεύουν οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και η σταθερότητα στην περιοχή. Γνήσια λύση στην, Κύπρο θα προέλθει, στην κρίση θα προέλθει μόνο από αμοιβαίο σεβασμό. Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ πρέπει να έχουν ως όρο το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Γι' αυτό ζητώ από Συμβούλιο και Κομισιόν να παγώσουν οποιαδήποτε αναβάθμιση των σχέσεων μέχρι η κατάσταση να έχει κάποια απτή βελτίωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Μάρικ Σίβιτς. Ευχαριστώ. Είμαι κατά των επικισμών, είμαι κατά των μονομερών κινήσεων. Αλλά αυτή είναι η πολιτική στην περιοχή μονομερείς κίνησει έχουν γίνει τόσο από τη μία όσο και από την άλλη πλευρά. Δυστυχώ έχουμε ακόμη και σήμερα να κάνουμε με αντιπαράθεση. Το Ισραήλ προβαίνει σε παρανομές κινήσει. Από την άλλη μεριά έχει να αντιμετωπίσει ρουκέτες. Και ο κόσμος τρέχει να κρυφτεί την τελευταία στιγμή. Μάνε με παιδιά έτρεχαν να κρυφτούν Όποιοι λοιπόν καταδικάζουν την επέκταση των οικισμών να θυμούνται ότι υπάρχουν δύο πλευρές σε κάθε νόμισμα. Ας είναι λοιπόν προσεκτικοί όταν καταδικάζουν. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν υπάρχει διάλογος, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για διάλογο. Το Ισραήλ παραμένει ακόμη εκτεθειμένο σε επιθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο ομιλητής, κυρία Μονίστα. Θα ήθελα να συγχαρώ το Συμβούλιο Ασφαλείας σε σχέση με την επέκταση των οικισμών του Ισραήλ. Καταδικάζουμε την επέκταση των οικισμών στη ζώνη ε1 που απειλεί ε, με μετακίνηση 2.300 Βεδουίνων. Επίσης, στη ζώνη ε, Γ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ως προς ε, σχέδια και υποδομές που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σχέδια που αφορούν την ηλιακή ενέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι όλες οι συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ θα πρέπει να παγώσουν τουλάχιστον στα κατεχόμενα. Και αυτό αφορά και την ε, Δυτική, Δυτική Όχθη και το Ανατολικό ε, Ισραήλ και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με Νομίζω ότι δεν είμαστε ε, διατεθειμένοι να απολέσουμε την Παλαιστίνη, να θυσιάσουμε την Παλαιστίνη όπως θέλουν μερικοί. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Σαρλάκη, πρόεδρε, η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι μετά τις εξελίξεις των ΟΗΕ θα συνεχίσει να επεκτείνει τους οικισμούς στην Δυτική Όχθη. Στέλνει έτσι το μήνυμα ότι δεν έχει κανένα σεβασμό για τα δικαιώματα του ανθρώπου και το διεθνές δίκαιο. Η κατασκευή των οικισμών αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Επιπλέον υπάρχουν νέα σχέδια για επικισμούς στη ζώνη ε1. Έτσι διακόπτεται η συνέχεια της δυτικής όχθης. Μειώνονται έτσι οι ελπίδες για ένα συνεχές αδιάλειπτο Παλαιστινιακό κράτος. Θυμίζω ότι το άρθρο 49 της Γενέβης απαγορεύει σε δυνάμεις κατοχής να καθιστούν πληθυσμό τους σε κατεχόμενες ζώνες. Γι' αυτόν τον λόγο υπογραμμίζω τη σημασία της δήλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία όλες οι συμφωνίες με το Ισραήλ πρέπει ρητός και περιφράστος να δηλώνουν ότι δεν εφαρμόζονται στα κατεχόμενα εκτός των συνόρων του Ισραήλ του 67 και δι στην Ρουρίδα της Γάζας, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Με εξέπληξε ο χαρακτήρας της σημερινής συζήτησης και οι τελευταίες συζητήσεις που είχαμε εδώ στο Κοινοβούλιο ως προς τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και Παλαιστίνης. Εμείς τασόμαστε υπέρ της ειρήνης. Το έχουμε εκφράσει ρητός και πάντα σεβόμασταν το κράτος του Ισραήλ. Ξέρουμε πόσες φορές ε, επαπειλήθηκε και απειλήθηκαν και οι υποδομές του, καθώς και οι πολίτες. Αλλά όταν αμφισβητούμε τις επισφαλείς αυτές σχέσεις και όταν απομακρύνεται η ειρήνη, τότε η κρίση μας θα πρέπει να είναι σαφής, δηλαδή να καταδικάσουμε τις πρόσφατες ενέργειες του Ισραήλ. Δεν μας βοηθά οποιασδήποτε αμφιβολία ως προς την ειρηνευτική αυτή διαδικασία. Η κυρία Μιράντα. Θα ήθελα να συγχαρώ την Παλαιστίνη για το νέο καθεστώς στο, στα Ηνωμένα Έθνη, το καθεστώς του κράτους παρατηρητή. Όμως οι επικισμοί είναι παράνομοι και αθέμητοι. Η έλεγχη, τα τείχη της ντροπή στα σπίτια τα οποία κλείνουν, τα εμπορικά καταστήματα που κλείνουν, το γεγονός ότι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν με ασφάλεια οι κάτοικοι μέσα στους επικισμούς, όλα αυτά μας αποθαρρύνουν. Η ασφάλεια είναι το πρώτο στο μέλημά μας και θα πρέπει να αποδώσουμε ένα σαφές μήνυμα προς την Ισραηλινή κοινότητα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αγκουράκης. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Αγκουράκης. Και αποχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρόταση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως κράτος παρατηρητή μη μέλους του ΟΗΕ αποτελεί ατράνταχτη απόδειξη του υπεριαλιστικού χαρακτήρα της πολιτικής και των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστινίους και τους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Το Ισραήλ εντείνει την επιθετικότητά του με απειλές για την κατασκευή τριών χιλιάδων κατοικίων για εγκατάσταση Ισραηλινών ε- επίκων στη ζώνη ανάμεσα στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως απάντηση στην πρόσφατη απόφαση του ΟΗΕ. Τώρα είναι επιτακτική η ανάγκη να εκφράσουν έμπρακτα οι λαοί την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό για ανεξάρτητο βιώσιμο κυρίαρχο Παλαιστινιακό κράτο στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, να σταματήσουν οι Ισραηλινοί επικισμοί στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και σε όλα τα Παλαιστινιακά εδάφη, συμπεριλαμβανομένων των υψωμάτων του Γκολάν και τη περιοχή Σεμπά στο νότιο Λίβανο, να αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός κατοχής και οι επίκη από όλα τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, την άρση κάθε αποκλεισμού της Παλαιστίνης, την άμεση απελευθέρωση όλων των Παλαιστινίων και την επιστροφή όλων των προσφύγων έτσι όπως ε, προτάσει ο Ευχαριστώ, Ιβο Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ότι γίνεται μια τέτοια συζήτηση ίσως δεν προσφέρεται για, προσωπικές τοποθετήσεις. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Έχω πάει κάποιες φορές στο Ισραήλ και πάντα είχα ως αφετηρία το ότι ήθελα να είμαι φίλος και των δύο πλευρών. Ίσως ε, να παίξω και ένα ρόλο μεσολαβητή. Θεωρώ πως ε, το βασικό πρόβλημα των σχέσεων Ισραήλ και Παλαιστίνης είναι η έλλειψη διαλόγου. Η έλλειψη επαφών των ανθρώπων και καλής θέλησης. Η σχέση λειτουργεί στο επίπεδο της ε, κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν θαυμάσιοι άνθρωποι οι οποίοι συνεννοούνται και μπορούν να ζήσουν το όραμα το οποίο περιέγραψε ο Άμος ως στο βιβλίο του ότι δηλαδή μπορούν να κάτσουν μαζί ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος και να πιούν έναν καφέ. Αυτή είναι η προοπτική. Νομίζω πως ε, το βασικό ελάττωμα της Ισραηλινής πολιτικής είναι πως ε, δεν θέλει να ε, ενδώσει σε αυτούς που βλέπουν το μέλλον, το αύριο και το μεθαύριο. Τέτοιο όραμα για το αύριο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ισραηλινή πολιτική. Ευχαριστώ. Κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώντας χρόνια όχι μόνο τα τραγικά γεγονότα αλλά και τις συζητήσεις πολιτικών από απόσταση και συχνά έτσι, κάπως αφηρημένα οι διάφορες ε, λύσεις και οι διατυπώσεις που χρησιμοποιούνται με ανησυχούν και θέλω να ρωτήσω όταν λέμε τόσα πράγματα για Παλαιστίνιους και Παλαιστίνοι ε, για ποια Παλαιστίνη και ποιους Παλαιστίνιους μιλάμε είναι υπάρχουν τουλάχιστον γεωγραφικά δύο Παλαιστίνες με δύο διαφορετικές δυνάμεις ή προσωπικότητες οι οποίες κυβερνούν. Το εάν ε, νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν ε, τμήματα του Παλαιστινιακού λαού είναι ένα ζήτημα. Αλλά ποιος εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους ε, πρόσφυγες. Ίσως πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι να γίνει μια αξιολόγηση. Να μην παίζουμε με τα λόγια Παλαιστίνη έτσι, η Παλαιστίνη έτσι, αλλιώ. Ποια Παλαιστίνη, η Παλαιστίνη της Χαμάς, του Αμπά είναι αναγνωρισμένη, η Χαμά αναγνωρίζει τον Αμπά ως νόμιμο πρόεδρο. Ας δούμε το ζήτημα ρεαλιστικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριος Μέρφυ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η εκπρόσωπος της ΕΠΑ της εκπροσώπου μας ενημέρωσε πως το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφές. Ας δούμε το μήνυμα της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δύο μήνες πέρασαν από όταν ψηφίσαμε να αναβαθμίσουμε τι εμπορικέ σχέσει με το Ισραήλ. Αύριο θα περάσουμε ένα ψήφισμα που θα ασκεί κριτική σε κάποιε πράξει του Ισραήλ. Το σαφέ μήνυμα νομίζω πω είναι το γνωστό. Προ την Ισραηλινή κυβέρνηση μην ανησυχείτε, λόγια μόνο λέμε, αλλά δεν θα κάνουμε ποτέ τίποτα και δεν αρκεί. Πρέπει άμεσα να ανασταλούν όλες οι συμφωνίες με το Ισραήλ. Με την οικοδόμηση των οικισμών γύρω-γύρω από την Ανατολική Ιερουσαλήμ κατ' ουσίαν ε, καταστρέφεται κάθε δυνατότητα βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους. Βλέπετε το τι σημαίνει λύση των δύο κρατών με βάση τον υπεριαλισμό και τον καπιταλισμό. Σημαίνει μπαντουστάν για τους Παλαιστίνιους θα υπάρξει μια μετεξέλιξη της Ιντιφάντας ή υποδημοκρατικό έλεγχο για να νικήσουν το δεξιό Ισραηλινό κατεστημένο και να συνδεθούν με τους εργαζόμενους όλου του κόσμου. Μόνο έτσι θα τελειώσει η καταπίεση των Παλαιστινίων και θα βρεθεί μια δίκαιη λύση με σοσιαλιστική Παλαιστίνη με ε, πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ δίπλα σε ένα σοσιαλιστικό Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριος Φαντάλεν. Ευχαριστώ. Πολλά ελέγχθησαν σήμερα, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Από την ημέρα της ύπαρξής του το Ισραήλ γνωρίζει τρομοκρατία και πόλεμο που δεν αναζήτησε το ίδιο το Ισραήλ. Και σήμερα η Χαμάς στην Δυτική Οχθή και στη Λωρίδα της Γάζας τρομοκρατεί το Ισραήλ. Αυτό δεν είναι καλό για τους ε, Παλαιστινίους. Τι μπορεί να κάνει το Ισραήλ από τον αντιδράσει. Δεν πιστεύω ότι οι, νέες, οι νέοι οικισμοί είναι η σωστή λύση, αλλά αυτό που θα πρέπει να επιδιώξουμε είναι να πούμε στη Χαμάς σταματήστε αυτή την τρομοκρατία τώρα. Αναγνωρίστε στο Ισραήλ και καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Παλαιστινιακή Αρχή. Αυτό θα πρέπει να ανακοινώσουμε στη Χαμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι οι νέοι οικισμοί δεν γίνονται σε καινούριο έδαφος, γίνονται σε έδαφος το οποίο είχε συμφωνηθεί, ήταν στο ε, territorial swap που υπάρχει συμφωνία από τότε με τον πρόεδρο Κλίντον δεν είναι λοιπόν κάτι καινούριο και κάτι παράνομο και θα ήθελα να απευθυνθώ στο κοινοβούλιο θα πρέπει να βλέπουμε με κάποια νυφαλιότητα την πολιτική αντίδραση του ισραήλ. το ισραήλ με την κίνησή του αυτή θέλει να υπενθυμίσει στην παλαιστίνη ότι ο διάλογος δεν έχει σταματήσει και πρέπει να συνεχιστεί και θα έλεγα προς όλους μας καλύτερα θα ήταν να ασχοληθούμε και να μας ανησυχεί η διαμάχη μεταξύ χαμάς και φατάχ παρά το γεγονός ότι το ισραήλ πράγματι αντέδρασε έτσι όπως έπρεπε να ε, κάνει για να στείλει ένα μήνυμα ότι ο διάλογος ακόμα συνεχίζεται. Ευχαριστώ κύριος Ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να μιλήσω. Ο κύριος Μέρφυ φεύγει. Ε, Αλλά αυτός με έκανε να μιλήσω γιατί ξέρω πως ε, παρακολουθεί πάρα πολύ τα ζητήματα του Καζακστάν. Εκτιμώ βεβαίως τη δραστηριότητά του αν και δεν συμφωνώ με την ιδεολογία του. Ξέρω πώς σας απασχολούν ζητήματα παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ασία. Αλλά γιατί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο κατά του Ισραήλ. Αυτό το φαινόμενο το παρατηρούμε εδώ και καιρό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιεβραϊκή, είναι κατά του Ισραήλ ε, με μια αριστερή έτσι, προσέγγιση. Όλα τα στραβά της Μέσης Ανατολής ε, τα κάνει το Ισραήλ. Ε, η κριτική της ε, αριστεράς είναι άνηση. Ε, Mr. Brock, you have the floor. Κύριος Μπρόκ έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Μα με προκαλεί αυτή η παρατήρηση από την άκρα αριστερά. Είναι σαφές πως θέλουμε μια λύση με δύο κράτη με βάση τα σύνορα του 1967. Πρέπει να υπάρχει ένα, μια βιώσιμη Παλαιστίνη και ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ. Πρέπει αυτό να γίνει γρήγορα και βεβαίως να υπάρξουν συνομιλίες. Αλλά να απαιτούμε σοσιαλιστική Παλαιστίνη και ότι αυτή είναι η μόνη λύση όταν η Χαμάς την τελευταία εβδομάδα ζήτησε να ε, καταπιεί ένα σεισμός το Ισραήλ και να εξαφανιστεί από τη γη. Ε, τι είναι αυτό, σοσιαλισμός, να εξαφανιστεί ένας λαός από το πρόσωπο της γης. Τελειώστε επιτέλους με το κομμουνιστικό σας μίσο, κα, μίσος κατά οποιοδήποτε δεν είναι ε, σοσιαλιστής. Δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να σταματήσουν κάποτε και αυτές οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Point of order, yes. But Επί διαδικασίας, αλλά να είναι επί της διαδικασίας. Και ορισμένοι άλλοι κύριοι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους και φεύγουν από την σκληρή πραγματικότητα που βιώνει καθημερινά ο Παλαιστινιακός λαός. Οι δολοφονικές επιθέσεις του Ισραήλ και η γενοκτονία ενάντια στον Παλαιστινιακό λαό είναι γεγονός I have the impression that it is not a point of order. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι επί της διαδικασίας αυτό. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη θέση ότι στη Μέση Ανατολή μπορούν να επιβιώσουν και οι δύο λαοί ως πλήρη ανεξάρτητα Λοιπόν, να σταματήσουν αυτές κορώνες εδώ και τώρα. Thank you. Thank you, please. Please. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Σας παρακαλώ ολοκληρώστε. Ναι, αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι τώρα η συζήτηση είχε μείνει εντός α, θέματος. Νομίζω πως ολοκληρώθηκε ούτως ή άλλως και θα ζητήσω από το Συμβούλιο να συνοψίσει ε, την στήριξη και την κριτική που ακούστηκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών τα συμπεράσματα είναι πολύ ε, στεναρά και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Μαζί με τα συμπεράσματα του Μαΐου του 2012 αποστέλουν ένα στεναρό μήνυμα σε όλους τους πρωταγωνιστές στον εδαφικό αυτό χώρο σε σχέση με την επίλυση του, ε, της σύραξης αυτής μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ. Είναι σαφέστατη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό δεν θα την επαναλάβω εμπεριέχεται στα συμπεράσματα που προανέφερα. Πρώτη στο μέλημα είναι να υποστηρίξουμε την ειρήνη και τη δημοκρατία σε ολόκληρη την περιοχή και στρατηγική μας προτεραιότητα είναι να σταματήσει αυτή η μακροχρόνια και τραγική σύραξη η οποία ε, υποδαβλίζει ε, υπονομεύει, με συγχωρείτε, την ειρήνη τη στιγμή που το ζήτημα αυτό δεν επιλύεται. Δεν θα υπάρξει βιώσιμη η ειρήνη εάν δεν δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος. Και παράλληλα το Ισραήλ θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένη την δυνατότητα ασφάλειας με βάση την λύση δύο κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει τα όσα προανέφερε στις 29 Νοεμβρίου στους Προέδρους Νεκτανιάχου και Αμπάς να συνεργαστούν για την επίλυση της ε, σύραξης αυτής και να δώσουν μια ε, νέα όθηση στις διαπραγματεύσεις μίλησαν ότι αποδέχονται τις άμεσες διαπραγματεύσεις χωρίς όρους. Προτρέπουμε και τις δύο πλευρές να το πράξουν και θα συνεργαστούμε μαζί τους. Μέσω ενός κουαρτέτου με την ε, συμμετοχή και τον ΙΠΑ, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μία βιώσιμη επίλυση του ζητήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες πρότειναν μία δήλωση η οποία θα συζητηθεί ή θα ψηφιστεί αύριο. Κλείνει η συζήτηση, θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι για το θέμα αυτό. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη εξ ονόματος της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και της ΥΠΑ της εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα